Madame la Présidente, mes chers collègues. Καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Επαναλαμβάνει τη συνεδρίαση. Μία ανακοίνωση. Τα συνοπτικά πρακτικά τη χθεσινής συνεδρίασης και τα κείμενα που εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση αυτή έχουν διανεμηθεί. Υπάρχουν παρατηρήσει. Δεν βλέπω κανέναν. Τα συνοπτικά πρακτικά λοιπόν εγκρίνονται. Το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι η έκθεση